πλέον σημαντική. Εδώ. Την έκθεση την αναβάλαμε ήδη μία φορά, γιατί μεταξύ εισηγητών υπήρξαν κάποιες ανάγκες συνεννόησης. Η σκιώδης εισηγήτρια των φιλελευθέρων δεν κατέθεσε τροπολογία τώρα έχει κάποια προβλήματα. Κυρία Σάκε, ακούστε τώρα που μιλάμε. Είναι ευγενικό να με κοιτάτε κιόλα, να μην φλιαρείτε την ώρα που μιλάμε για σας. Θα εγκρίνουμε μία έκθεση λοιπόν που είχε αναβληθεί λόγω διαφορετικών απόψεων. Και τώρα ανεξάρτητα από κάθε προθεσμία. Έχουμε εδώ τη λεγόμενη ψήφο μειοψηφία που πρέπει να την δεχτούμε ε, είτε θέλουμε είτε όχι, ε, συνημένη στην αιτιολογική έκθεση της κυρίας Κώστα. 23 χρόνια είμαι ευρωβουλευτής και τέτοιο πράγμα δεν ξανάδα. Είναι τελείως άδικο η κυρία Σάκε δεν κατέθεσε ούτε μία τροπολογία. Άρα δεν συμμετείχε στις προετοιμασίες και έρχεται μια μέρα πριν από την ε, ψηφοφορία που ήδη είχε αναβληθεί με ψήφο μειοψηφίας. Είναι πολύ άδικο αυτό και απέναντι στην συνάδελφο εισηγήτρια και απέναντι σε όλους μας. Η δουλειά κυρία Σάκε γίνεται εδώ κατά τις συζητήσεις. Εσείς δεν κάνατε ούτε μία τροπολογία. Τέτοιο πράγμα δεν μου συνέβη ποτέ τόσα χρόνια και νομίζω ότι δεν είναι ευγενικό απέναντι στους συναδέλφους. Δυστυχώς είμαι υποχρεωμένη να το δεχτώ ως διαδικασία γιατί προβλέπεται από το καταστατικό. Μπορεί όλοι να λέμε ότι είναι άδικο, αλλά δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει λοιπόν να μπει στα πρακτικά μας τη συνεδρίασης ότι αυτό είναι άδικο και αντισυναδελφικό απέναντι σε όλα τα μέλη της Επιτροπής. Και επί της ουσίας ε, δεν στέκει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Επαναλαμβάνω, Είμαι 37 χρόνια βουλευτής, τέτοια, ε, είμαι βουλευτής 37 χρόνια. Τέτοια συμπεριφορά δεν είδα από κανέναν και θέλω να γραφτεί στα πρακτικά παρακαλώ. Λοιπόν, ευτυχώς ε, Σίλβια τα φέραμε εις πέρας όλα αυτά. Έχεις το λόγο για να μας ε, πεις. Και ελπίζω κύριε Στάκουλα να ντρέπετε. Κυρία Κώστα. Grazie, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Νομίζω ότι είπατε και σας ευχαριστώ για αυτά που είπατε και με τη δέουσα αυστηρότητα που έχει και σχέση για το fair play που πρέπει να υπάρχει μεταξύ των συναδέλφων σε αυτήν την Επιτροπή. Απλώς να πω, θα ήθελα, δεν θα προσθέσω τίποτε άλλο, ότι πραγματικά με ξένησε, με εντυπωσίασε αυτή η συμπεριφορά. Γιατί έφτασε χθε το βράδυ στις 8.30 από την εισηγήτρια του Άλτα δεν είχα πάρει καμία τροπολογία, εργαστήκαμε βάσει των τροπολογιών της συναδέλφου Ήρσου της ομάδος και μου φαίνεται ότι κάναμε τελικά με ένα λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα μια γνωμοδότηση η οποία πιστεύω πως σε τελική ανάλυση προσπαθεί να ερμηνεύσει τις απαιτήσει πολλών συναδέλφων πραγματιώντα πολλούς συμβασμού. Αυτό ήθελα να πω, δεν θα να προσθέσω τίποτα άλλο σε αυτά που είπατε. Λυπούμε. Ελπίζω να το ξανασκεφτεί για να το ξανασκεφτούν αυτοί οι συνάδελφοι. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη γνωμοδότηση αυτή, να ευχαριστήσω όλου που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στην επεξεργασία αυτή, τη Γραμματεία βεβαίω για την στήριξη την οποία μου προσέφερα και τη Στεφανή ειδικότερα, και κυρίω διότι πιστεύω ότι σε επίπεδο και σε ένα θέμα τόσο λεπτό και ευαίσθητο όπω είναι η προστασία των ανηλίκων, τόσο για να προωθηθεί η δική του ενεργό συμμετοχή στον ψηφιακό κόσμο, όπω επίση και για να προστατευτεί η αξιοπρέπεια αυτών και η δυνατότητα να μπορούν να έχουν προσχώρηση και να προσβάσουν πρόσβαση σε ένα δίκτυο πιο ασφαλές στο διαδίκτυο δηλαδή, νομίζω ότι κάναμε καλά, καλή δουλειά και ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Αρχίζουμε λοιπόν την ψηφοφορία. Τροπολογία 65 υπέρ. Παρέμβαση εκτός μικροφώνου. Ψηφίζουμε. Δεν σας γνωρίζω κύριε, δεν σας έχω ξαναδεί στα μάτια μου, αλλά ψηφίζουμε αυτή τη στιγμή. Και έχω εγώ το λόγο. Εφόσον είστε στην Επιτροπή Πολιτισμού, να έρθετε στην ώρα σας, όπως και εγώ. Τώρα εγώ έχω το λόγο, η ψηφοφορία ξεκίνησε. Αρχίζουμε με την τροπολογία 65. Ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 65. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 73. Υπέρ. Κατά. 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 72. Όχι, 75. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 76 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά αποχές θα το ελέγξουμε αυτό. Άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία 78. Πέρα της ψηφοφορίας. 14 προς 13 υπέρ. 70 υπέρ. Κατά αποχές Όχι, 70 καταπίπτει. Πάμε στη συμβιβαστική 2. πάμε ή δεν πάμε στη συμβιβαστική 2. Ναι, συμβιβαστική 2 λοιπόν. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 83 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 84 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 85 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε. 88. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 16 προς 12 εγκρίνεται. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ελέγχουμε την 89. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 13 προς 15 απορρίπτεται. Συμβιβαστική 3. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην 96. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 98 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 99 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 100 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 102 υπέρ. Κατά αποχές έλεγχος. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουμε την 102. Πέρας. 15 προς 13 απορρίπτεται, 103 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 110 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές δεκτή 113 υπέρ Α, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Την 110 θα ψηφίσουμε, όλα τα άλλα καταπίπτουν. 116 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 117 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή, 118 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές δεκτή 120 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ Α, είχε γίνει ήδη δεκτή. 123. Έμα Μακλάρκιν, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 131 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 132 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 133 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 134 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 135 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 137 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 138 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 139 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 140 υπέρ κατά αποχές δεκτή 141 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 142 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 143 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται 144 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 145 υπέρ, κατά αποχές δεκτή 146 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 152 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 153 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 154 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 155 υπέρ κατά αποχές απο, ε, δεκτή, 156 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 157 υπέρ κατά αποχές έλεγχος, 157 ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 15 προς 13 δεκτή, 158 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 160 υπέρ κατά αποχές δεκτή 161 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 162 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία την 164 πέρας 17 προς 10 δεκτή. 165 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 166, 167 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 168 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 169 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 170 υπέρ κατά αποχές δεκτή 171 υπέρ κατά αποχές δεκτή 172 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή 174 υπέρ κατά αποχές δεκτή 173 υπέρ α, με συγχωρείτε λέει πρόεδρος 176 φωντάνα υπέρ κατά αποχές έλεγχος στην 176 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. 17 προς 11 δεκτή. 177 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 178 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 179 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 180 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 182 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές, έλεγχος, άρχεται η ψηφοφορία, στο τροπολογία 11. Πέρας. 16 προς 10 απορρίπτεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Όχι, ε, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Στην 20 θα ψηφίσουμε τώρα. 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 23 υπέρ κατά αποχές δεκτή 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 όχι ε, ναι, 28 ε, όχι, ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, τμήματική ψηφοφορία στην 29. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. 30 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 11. 7 ε, συγγνώμη υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 37 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 38 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ. Όχι, 43. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε λέει η πρόεδρος. Τη 43 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή 55 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 57 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 59 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 60 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 61 υπέρ κατά αποχές δεκτή 62 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές δεκτό. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Πάμε τώρα στην λίμπε 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Λίμπε 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή, η 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικά θα γίνει. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 20 υπέρ 3 κατά 4 αποχές δεκτή. Ε, συγχαρητήρια θερμά κυρία Ντακώστα. Ευχαριστώ σε όλους, ευχαριστώ και την Προεδρία. So we come to the next... Και προχωρούμε στην επόμενη έκθεση. στο σημείο 8 της ημερήσιας διάταξης. Η έκθεση του κυρίου Μπόρις για την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Κύριε Μπόρις, έχετε το λόγο για να μας παρουσιάσετε τις σκέψεις σας και τις ιδέες σας. Ορίστε. E, dziękuję bardzo. E, szanowne panie, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίε και κύριοι, μέλη τη Επιτροπή. Πρόκειται για την πρώτη ανταλλαγή απόψεων σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων. Είναι μία από τις πλέον σημαντικές νομοθετικές πράξεις πάνω στις οποίες, στην οποία μάλλον έχει εργαστεί η δική μας Επιτροπή επί σειρά ετών. Θα ήθελα να θυμίσω σε όλους, ο, η τελευταία αναθεώρηση της οδηγίας αυτής πραγματοποιήθηκε μεταξύ του 2005 και του 2007. Και αυτό που συνέβη ήταν η σύγκληση όλων των οπτικοακουστικών μέσων και η μετάδοση του οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω Ενό μεγαλύτερου αριθμού από πλατφόρμες. Σκοπός της οδηγίας αυτού ήταν η εισαγωγή των μη γραμμικών αποβαλμένων υπηρεσιών. Και να ρωτήσω τώρα, αν μου επιτρέπετε, το γιατί πρέπει να συζητήσουμε και θέλουμε να συζητήσουμε την έκθεση αυτή, διότι το άρθρο 33 καθιστά δυνατόν να αξιολογήσουμε και να αξιολογηθεί η εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Δυστυχώς η έκθεση αυτή έχει καθυστερήσει κατά περίπου μισό έτος, διότι δεν ήταν στη θέση όλα τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν, να υλοποιήσουν την οδηγία αυτή. Διότι μόνο 23 κράτη-μέλη υλοποίησαν την οδηγία αυτή. Τα άλλα τέσσερα κράτη-μέλη βρίσκονται καθοδόν, αλλά συναντούν κάποιες δυσκολίες, ειδικότερα το Βέλγιο και η Πολωνία, με την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Οι διαπραγματεύσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχουν ξεκινήσει και νομίζω πω η διαδικασία αυτή θα κλείσει, θα οριστικοποιηθεί σχετικά σύντομα. Νομίζω ότι έχουμε και θα έχουμε ένα πολύ σημαντικό και πολύτιμο εργαλείο στα χέρια μα. Διότι η διηγία αυτή εστιάζεται σε δύο σημεία, σε δύο στοιχεία. Την υλοποίηση, την εφαρμογή του, των κανονισμών που αποσκοπούν στην προστασία των ανηλίκων που ήταν ένα από του στόχου αυτή τη οδηγία ό,τι αφορά τι υπηρεσίε οπτικοακουστικών μέσων. Η πρόσβαση στην πληροφορία ήταν επίση ένα άλλο πολύ σημαντικό σημείο, αλλά ένα πολύ σημαντικό σημείο από τη δική μα σκοπιά είναι ότι όλα αυτέ οι προσπάθειε θα γίνουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο δεύτερο κομμάτι τη έκθεσή μου ασχολούμαι με την αξιολόγηση τη οδηγία ειδικότερα σε ό,τι αφορά τις τα νέα σημεία των ε, οπτικοακουστικών υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, τα μη γραμμικών. Στο πλαίσιο της υβριδικής αποκαλούμενης τηλεόρασης, όπως επίσης και στο πλαίσιο ε, των προκλήσεων της, ε, της σημερινής κατάστασης. Αλλά όχι μόνο οι μη γραμμικές υπηρεσίες, αλλά και άλλες υπηρεσίες που έχουν σχέση με την πρόσβαση ή το περιεχόμενο καταζήτηση, το on demand. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να πω είναι ότι θέλουμε να αξιολογήσουμε θετικά την οδηγία αυτή. Διότι πιστεύω ότι η οδηγία αυτή φέρνει επανάσταση έτσι ώστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε ελεύθερη κυκλοφορία οπτικοακουστικού περιεχομένου και ω προ αυτό υπήρξαμε αρκετά επιτυχεί κυρίε και κύριοι, διότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι σήμερα οι εταιρείε παραγωγή μπορούν να απολαύουν τις ελευθερίες των. Δεν χρειάζονται ειδικέ και ιδιαίτερε άδειε για προκειμένου να εκπέμπουν και να μεταδίδουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Σε ό,τι αφορά την ελευθερία κίνηση, η οδηγία αυτή πραγματικά έχει αποδείξει την αξία της. Να πω λίγα λόγια τώρα, αν μου επιτρέπετε, για την εφαρμογή, την υλοποίηση κάποιων διατάξεων που αφορούν στην προστασία των παιδιών, των ανηλίκων. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να επισημάνω και να τονίσω κάποια συμπεράσματα τα οποία μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η ελευθερία και ο πλουραλισμός στα μέσα έχουν διατηρηθεί. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω επίσης θα ήθελα και ότι σε ό,τι αφορά την προστασία σε σχέση με την, από τη μυσαλλοδοξία που ήταν τα βασικά στοιχεία που αποσκοπούσαν στην προστασία των ανηλίκων ως προς αυτό το σημείο η οδηγία λειτουργεί πολύ καλά μάλιστα. είχαμε ένα επεισόδιο στη Γαλλία όταν ένα από τα κανάλια μετέδωσε κάποια, κάποια αντισημιτικά μηνύματα, αντισημιτικό περιεχόμενο. μέσω του Utelsat, του δορυφόρου. Και το περιεχόμενο αυτό δεν κατέστη διαθέσιμο. Πράγμα το οποίο δείχνει πόσο επιτυχής υπήρξε η οδηγία αυτή και ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο, σε παράδειγμα, τι θα ήθελα να πω, ότι η οδηγία πραγματικά αποδίδει καρπού σε ό,τι αφορά την προστασία των νέων. Προστασία των νέων από επικίνδυνο περιεχόμενο. Τώρα, α περάσουμε στο ζήτημα της πρόσβασης σε οπτικοκουστικό περιεχόμενο. Ως προς αυτό παρατηρήσαμε ότι υπήρξε βελτίωση, σημειώθηκε βελτίωση. Ειδικότερα σε εκείνους που έχουν προβλήματα είτε όρασης είτε ακοής. Τώρα είναι σε καλύτερη και πολύ καλύτερη θέση και έχουν πρόσβαση σε αρκετό οπτικοκουστικό περιεχόμενο. Πολύ περισσότερο από στο παρελθόν. Ωστόσο προ αυτό το σημείο δηλαδή η λειτουργία λειτουργήσε αρκετά καλά. Η οδηγία αυτή επίση προσφέρει κατοχυρώνει κάποια δικαιώματα, για να το θέσω διαφορετικά, σε ό,τι αφορά την πρόσβαση σε συγκεκριμένο περιεχόμενο. Φερρυπίν. Υπάρχει ένα περιεχόμενο κοινωνικό σοβαρό, το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία για πολλά κράτη-μέλη. Φερρυπίν, αθλητικές εκδηλώσει είναι επίση πολύ σημαντικέ και έχουν σχέση βεβαίω και με τι εργασίε τη δική μα Επιτροπή, διότι στο Βέλγιο και στο Ηνωμένο Βασίλειο αποφασίστηκε ότι τα δικαιώματα εκπομπής και αναμετάδοσης αγώνων ποδοσφαίρου στο πλαίσιο της FIFA ή της UEFA θα πρέπει να είναι προσπελάσιμε από όλους. Και αυτό εγγράφεται και στο πλαίσιο του καταλόγου που διατέθη σε όλους. Ένα επιθυμητό περιεχόμενο δηλαδή για όλους τους ε, θεατές, τηλεθεατές και ακροατές βεβαίως ελήφθησαν υπόψη όλε οι τυχέ τη κοινωνική ζωή. Και υποχρεωτικώ θα πρέπει να διαθέσουμε αυτό το περιεχόμενο σε όλου. Σε ό,τι αφορά τώρα τι εργασίε τη δική μα επιτροπή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η οδηγία αυτή λειτουργήσε αρκετά καλά. Και αναφέρομαι εδώ στην πολιτισμική ισότητα που πρέπει να υπάρχει. Η οδηγία έχει διατάξει που αφορούν κάποια, σε κάποια ελάχιστα όρια που σχετίζονται, συνδέονται με την εκπομπή και προγραμμάτων στην Ευρώπη. Να πω επίσης θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, ότι για τους σκοπούς της προώθησης του πολιτιστικού περιεχομένου η οδηγία αυτή από αυτή την πλευρά λειτουργεί πολύ καλά. Οι εταιρείε θα πρέπει ένα συγκεκριμένο ποσοστό των εκπομπών που θέλουν να κάνουν στην Ευρώπη θα πρέπει να το διαθέσουν σε ανεξάρτητες εταιρείε. Παρακολουθώντας βεβαίω και το πώς γίνονται αυτές οι εκπομπές σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συν πλην 62% μέχρι το 2008. Αλλά σε ό,τι αφορά τις ανεξάρτητες αυτές εκπομπές 35%. Η οδηγία αυτή μας έδωσε ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να εισάγουμε και να θεσπίσουμε μια ελάχιστη ποσόστοση για ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκά προγράμματα και για την εκπομπή αυτών και την αναμετάδοσή των. Το ποσοστά αυτά νομίζω ότι είναι αρκετά λογικά. Και ποιο είναι το συμπέρασμα, ότι μπορέσαμε με τον τρόπο αυτό να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή αγορά πολιτιστικού περιεχομένου και έργων πολιτισμού. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα ήθελα, στο να αναφερθώ είναι και το ζήτημα των διαφημίσεων, των τηλεοπτικών, σποτ και άλλων. Η οδηγία αυτή ορίζει σαφώς το τι συνιστά τηλεοπτικό σποτ. Και ξέρουμε βεβαίως πόσο δύσκολο είναι να προστατευτούν οι καταναλωτές έναντι κάποιων τάσεων που αρχίζουν να διαμορφώνονται στον κόσμο της τηλεόρασης να χρησιμοποιούνται πολύ έντονα και εντατικά οι τηλεοπτικές διαφημίσεις. Πολύ συχνά όταν παρακολουθούμε μια ταινία φερειπίνη στην ε, τηλεόραση υπάρχουν πολλά διαλύματα κατά διάρκεια των οποίων μεταδίδονται πολλά, ε, πολλές διαφημίσεις. 12 λεπτά διαφημίσουν σε μια εκπομπή 60 λεπτών, σε ένα πρόγραμμα 60 λεπτών. Αυτή είναι η τακτική η οποία έχει υιοθετηθεί και ακολουθείται. Αλλά στα περισσότερα κράτη-μέλη τα όρια αυτά έχουν δυστυχώ παραβιαστεί. Η τηλεόραση δηλαδή προχωράει προσπαθεί, προσπαθώντας βεβαίως να γεφυρώσει το χάσμα που υπάρχει. Το ζήτημα της προστασίας των θεατών έναντι υπερβολικών ε, διαφημιστικών μηνυμάτων δεν είναι κάτι το απολύτως ε, εξασφαλισμένο. Γιατί αυτό το όριο που υπάρχει έχει παραβιαστεί από πολλές διαφημιστικές εταιρείες. Βεβαίως ε, εφαρμόζονται και προσπαθούνται πολλές ε, μέθοδοι προκειμένου να υπερβαθεί αυτό το όριο των 12 λεπτών διαφημίσεων σε διάρκεια ενός 60 λεπτού προγράμματος. Να μιλήσω τώρα για την ισότητα. Έχουμε κάποια εργαλεία, η οδηγία δηλαδή έχει κάποια εργαλεία που σκοπό έχουν να προστατεύσουν τα παιδιά έναντι υπερβολικών διαφημίσεων τηλεοπτικών. Και υπάρχει και ένα εργαλείο με το οποίο μπορούμε να παρακολουθήσουμε και να επιτηρήσουμε την κατάσταση. ε, διαφημίσεις για το αλκοόλ, για ενοπνευματόδη ποτά, που πολλές φορές φτάνουν και το 3% του τηλεοπτικού χρόνου. από 3 8%. Αλλά έχουμε επίσης και ένα άλλο τμήμα στην οδηγία, το οποίο μας προστατεύει από κάποια τηλεοπτικά σποτ που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνα για τα παιδιά νεαρότερης ηλικία. Περιπίν σε πέντε κράτη-μέλη, Φερρυπίν σε κράτη-μέλη, απαγορεύεται η αναμετάδοση διαφημίσεων κατά τη διάρκεια προβολής προγραμμάτων για τα παιδιά. Αυτό είναι ο λόγο για τον οποίο εν γέννη θα μπορούσα να πω ότι η οδηγία και με τρόπο αποτελεσματικό μάλιστα προστατεύει τα παιδιά απέναντι σε ανεπιθύμητο περιεχόμενο. Διότι τα παιδιά είναι και τα πιο ευάλωτα και θα μπορούσαν πολύ περισσότερο από ότι οι μεγαλύτεροι να επηρεαστούν από το περιεχόμενο αυτό. Και νομίζω πως η οδηγία αυτή τελικώς έχει εξυπηρετήσει το σκοπό και οι τρόποι προστασίας των παιδιών από τέτοιου είδους διαφημίσεις και τηλεοπτικά σποτ είναι καλή. Να πω τώρα κάτι το οποίο είναι λεπτό και ευαίσθητο ζήτημα από, όπως προκύπτει την ανάλυση αυτών των τηλεπτικών σποτ είναι ότι οι στερεότυπες ε, στάσεις σε ό,τι αφορά το φύλλο ε, ύψιλον την εθνικότητα διαπλέκονται στο 20 30% των ε, διαφημίσεων. Οι διαφημίσεις βεβαίως βασίζονται σε κάποια στερεότυπα γιατί μπορούν να φτάσουν και θέλουν να φτάσουν στο μυαλό των θεατών πιο αποτελεσματικό τρόπο και να μπουν μέσα σε αυτό, για να το θέσω απλά. Ε, από αυτή την έννοια η οδηγία θα μπορούσε να εξυπηρετήσει και να παίξει το ρόλο ενός αστυνόμου, ο οποίος συνεχίζει και συνεχώς μας υπενθυμίζει τι είναι νόμιμο και τι όχι, τι μπορούμε να κάνουμε και τι όχι. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε να επιτηρούμε, να παρακολουθούμε την κατάσταση, διότι τα στερεότυπα στις διαφημίσεις πολύ συχνά χρησιμοποιούνται. Πιστεύω ότι η οδηγία αυτή εκπληρεί τον στόχο της, προστατεύει δηλαδή τον θεατή, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την εφαρμογή της. Η αυτορύθμιση είναι επίσης ένα άλλο πολύ σημαντικό στοιχείο της οδηγίας αυτής, διότι υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να προστατεύσουμε τους τηλεθεατές και ειδικότερα τους νεαρούς, τους νέους, μικρή της ηλικία από διαφημίσεις με περιεχόμενο που σχετίζεται Φερρυπίν με την υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρές ή σε ζάχαρα κάποιων ε, ειδών διατροφής. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταπολυθούν τα, οι διαφημίσει, οι τηλεοπτικέ διαφημίσει, οι οποίε δεν αρμόζουν στα παιδιά. Ειδικότερα σε αφορά τη, τα διάφορα τρόφιμα, οι διάφορα είδη διατροφή που διαφημίζονται. Η αξιολόγηση πάντω τη οδηγία, που έρχεται με καθυστέρηση 6 μηνών περίπου, σε ό,τι αφορά τον πλουραλισμό στα μέσα ενημέρωσης, και με σκοπό βεβαίως και την πρόθεση του ευρωπαϊκού οπτικοακουστικού περιεχομένου στα προγράμματα τα οποία μεταδίδονται στην Ευρώπη οδηγούν σε μια θετική αξιολόγηση. Τα εργαλεία τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιούμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να είναι τα σαφή μηνύματα που θα πρέπει να εκπέμπουμε διασφαλίζοντας βασικά στοιχεία της οδηγίας αυτής δεν βρήκα ως προς αυτό τίποτε το ονοχοποιητικό, τίποτε βεριπίν το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια πολύ σημαντική αναθεώρηση της οδηγίας αυτής. Βεβαίω τα κράτη-μέλη θα πρέπει να εφαρμόσουν έγκαιρα τα διάφορα στοιχεία και σημεία αυτής της οδηγία και εμεί να παρακολουθούμε βεβαίω και να επιτηρούμε για να ξέρουμε τι ακριβώ έχει συμβεί και τι συμβαίνει. Τώρα βεβαίω, ο αντίκτυπος της οδηγίας αυτής ε, σε ό,τι φορά τις νέες τεχνολογίες και εννοώ την υβριδική τηλεόραση την αποκαλούμενη είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Η οδηγία ή το τεχνολογικό σου δέτερη διότι οι διατάξεις της, της οδηγίας αυτής δηλαδή σχετίζονταν με κάθε είδους οπτικοακουστικής υπηρεσίας. Η συνάδελφος βεβαίως ετοιμάζει μια ιδιαίτερη έκθεση σε ό,τι αφορά την υβριδική αποκαλούμενη τηλεόραση και σήμερα αυτές οι γραμμικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται με τρόπο πιο περιοριστικό από τον νόμο. Οι μη γραμμικές υπηρεσίες αντιμετωπίζονται διαφορετικά. Αλλά συνεχίζω να πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε πείγνωση του γεγονότος ότι έχουμε να κάνουμε με δύο διαφορετικές πραγματικότητες την γραμμική και την μη γραμμική τηλεόραση. Τα προγράμματα των οποίων είναι πολύ διαφορετικά μεταξύ τους. Τα μη γραμμικά προγράμματα της μη γραμμικής τηλεόρασης αλλάζουν τώρα και δραματικά μάλιστα. Και νομίζω ότι προσπαθώντας να προστατεύσουμε και να προστατευτούμε από τα στοιχεία τα οποία σας περιέγραψα στην αρχή της παρουσίασής μου, πρέπει να δώσουμε στους εαυτούς μας μια πίσωση χρόνου, έτσι ώστε να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και να εφαρμόσουμε τις νέες τεχνολογίες, παρακολουθώντας πολύ προσεκτικά τις εξελίξεις της μη γραμμικής αποκαλούμενης τηλεόρασης, της υβριδικής τηλεόρασης και το πώς οι υπηρεσίες αυτές θα μπορούσαν και τι αντίκτυπο θα έχουν σε σχέση με την ε, υλοποίηση, την εφαρμογή, την εκτέλεση της οδηγίας. Ως προς αυτό νομίζω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει στα χέρια του πλέον ένα πολύ καλό μέσο και θα πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την υλοποίηση, την εφαρμογή της οδηγίας αυτής. Γενικώ πώς είναι πολύ καλή η οδηγία αυτή, αλλά το μόνο που χρειάζεται τώρα πλέον είναι να φροντίσουμε να εφαρμοστεί και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα σας παρουσιάσω νομίζω μια περαιτέρω έκθεση επί του αυτού αργότερα. Και βεβαίω τα σχόλια της παρατηρήσεις σα θα ήθελα να ακούσω σε σχέση με αυτά που σας παρουσίασα, με ενδιαφέρουν όλος ιδιαίτερος, γιατί νομίζω πως ε, πρέπει να έχουμε ένα ευρύ πεδίο συζήτηση όσον αφορά την υλοποίηση οδηγία και ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μπόρις για την ανασκόπηση που μας κάνατε. Η Πέτρα Κάμαρτε καταρχήν, μετά Έγραψα και εγώ τον, το όνομά μου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Πιότρ για την παρουσίαση της έκθεσής σου. Νομίζω ότι η έκθεση της Κομισιόν δείχνει σαφώς ότι τότε με την οδηγία από την τηλεόραση χωρίς σύνορα σε μια οδηγία, το πέρασμα σε μια οδηγία για, για τα οπτικοακουστικά εστιάσαμε στη, στα οπτικοακουστικά και αυτό ήταν σωστό. Βρήκαμε άλλωστε και το σωστό μέσον, ούτω ώστε να ρυθμιστούν σε πολιτικό επίπεδο αυτά που έπρεπε να ρυθμιστούν και αναδείξαμε και τον ιδιαίτερο χαρακτήρα των οπτικοακουστικών μέσων, τις ιδιαιτερότητες του σε σχέση με την εξέλιξη της κοινωνίας, τα μέσα, την ελευθερία της επικοινωνίας και της έκφρασης. Όλα αυτά λαμβάνονται υπόψη με όλος ιδιαίτερο τρόπο και θα πρέπει να διατηρήσουμε την οδηγία ε, λειτουργική και στο μέλλον. Συμφωνώ ότι η οδηγία σε μεγάλο βαθμό λειτουργεί, είναι αποτελεσματική. Πρέπει όμως να δούμε κυρίως το διαφημιστικό κομμάτι. Γιατί εκεί ότι υπάρχει μια, ένας δημιουργικός χειρισμός των κανόνων και μια ευρύτατη ερμηνεία. Πολλές φορές οι διαφημίσεις ε, ονομάζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να ξεφεύγουν από, τον κανόνε από τους κανόνες μας. Να δούμε, την, να δούμε την υβριδική τηλεόραση, τους κανόνες που έχουμε, για ποιους επιμέρους τομείς και σε ποια σημεία θα πρέπει να επιφέρουμε βελτιώσεις. Μια ιδιαίτερη πρόκληση θα είναι η ανάπτυξη καινούριων μορφών διαφήμισης, ακριβώς με κίνητρο να υπο ε, να, να, ξεφύγουν από τους κανόνες και αυτό θα πρέπει να το δούμε και σε σχέση με τη συνδεδεμένη τηλεόραση ή την υβριδική γιατί οι νέες τεχνολογίες ανοίγουν νέες δυνατότητες ε, αντιμετώπισης των, ε, και, και ανάμειξης των τηλεοπτικών ε, σημάτων. Είμαι πεπισμένη ότι στα πλαίσια της εξέλιξης της τεχνολογίας χρειαζόμαστε και επιμέρους ρυθμίσεις στα οπτικοακουστικά μέσα. Δεν μπορούμε δηλαδή να περάσουμε μια οδηγία ηλεκτρονικού εμπορίου και να ε, ρυθμίζουμε και αυτά τα θέματα σε σχέση με το δίκαιο ανταγωνισμού. Θα πρέπει να δούμε τον ειδικό χαρακτήρα των μέσων και να έχουμε μια ρύθμιση αποκλειστικά για αυτά. Στην έκθεσή μου για το Connected TV θα τα αναφέρω κι εγώ, διότι νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλές προκλήσεις που πρέπει να μας απασχολήσουν και μάλιστα πρέπει να δράσουμε και σχετικά γρήγορα για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις. Αλλιώς ε, υπάρχει ο κίνδυνος να ισχύσουν τα τετελεσμένα γεγονότα και ε, να έχουμε κάποιες ε, επιχειρηματικές κινήσεις που θα εξελιχθούν και θα παγιωθούν και μετά θα τις δούμε εμείς. Οπότε θα είναι ίσως πολύ αργά για να αντιδράσουμε. Πρέπει λοιπόν έγκαιρα να κάνουμε κάποιες σκέψεις για να δούμε πώς την ε, ε, σχετική οδηγία να την επεκτείνουμε για να συμπεριλάβει τη συνδεδεμένη τηλεόραση, Connected TV και να ε, παραμείνουν διασφαλισμένες η προστασία των νέων, ε, η ενότητα κάποιων, η χαρακτήρας κάποιων κανόνων για τις διαφημίσεις κλπ. Όλα αυτά θα είναι μια μεγάλη πρόκληση και είπα ήδη ότι πρέπει να δράσουμε έγκαιρα ούτως ώστε να δράσουμε προληπτικά πριν μας ξεπεράσουν οι εξελίξεις. Ε, στην παρουσίαση της έκθεσης η κυρία Κώστα είπε πολύ... Ε, ε, ο εισηγητής είπε ότι η οδηγία ε, λειτουργεί ως έχει, αλλά παράλληλα είπε ότι πρέπει να παραμείνουμε στο παιχνίδι και να λάβουμε υπόψη μας και όλες τις εξελίξεις στα πλαίσια του Connected TV. Η ΔΕ Κομισιόν είπε ότι θα αρχίσει μια διαδικασία διαβουλεύσεων και νομίζω και η έκθεση πρωτοβουλίας που ετοιμάζω εγώ θα είναι μια συμβολή σε αυτή τη διαδικασία συμβούλευσης όπου και εμείς ως Κοινοβούλιο έγκαιρα θα μπούμε στη συζήτηση για τις ρυθμιστικές ανάγκες του Connected TV. Ε, έτσι πιστεύω ότι η έκθεση για την ε, ε, εφαρμογή της οδηγίας για τα οπτικοακουστικά και η δική μου έκθεση θα μπορέσουν να αλληλοσυμπληρωθούν με πολύ θετικό τρόπο και περιμένω και στο μέλλον να έχουμε πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Ευχαριστώ λοιπόν την Πέτρα, ευχαριστώ τον κύριο Μπόρις. Θυμάμαι όταν κάναμε διαβουλεύσεις για την οδηγία και λέγαμε αφενός ότι θέλουμε τον προσανατολισμό προς την εσωτερική αγορά και να περάσουμε από την έννοια της τηλεόρασης στην έννοια των οπτικοακουστικών γιατί θέλουμε να συμβαδίσουμε με τους καιρούς και πρέπει κιόλας και παράλληλα με τον προσανατολισμό ε, της εσωτερικής αγοράς λάβαμε υπόψη και το διασυνοριακό χαρακτήρα και θέλαμε να περιορίσουμε τις διαφημίσεις με κανόνες. Ε, σε ό,τι αφορά την υποκίνηση σε μίσος, τις ρυθμίσεις για τις διαφημίσεις, ε, όλα αυτά λοιπόν που έχουν να κάνουν με την εσωτερική αγορά και το διασυνοριακό της χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη ε, θέματα πολιτισμικά και οικονομικά εμπορικά. Τώρα, κάποια σχόλια πάνω σε αυτά που ακούσαμε. Γενικά συμφωνώ με την προσέγγιση της Πέτρας ε, ότι θα πρέπει η οδηγία να παραμείνει λειτουργική. Δεν είναι λάθος, ούτε είναι τελείως ξεπερασμένη, αλλά θα πρέπει να προσαρμοστεί. Πιστεύω ότι η έκθεση πρωτοβουλίας για το Connect TV και τι γίνεται με τις μη γραμμικές προσφορές και όλες τις προσφορές μέσω διαδικτύου, να τα δούμε αυτά, και τις γραμμικές ε, προσφορές, όλα αυτά θα πρέπει να τα δούμε από κοινού και να τα εξετάσουμε στην Επιτροπή. Δεν μπορούμε να διαχωρίσουμε πια τους δύο κόσμους, άρα ούτε οι δύο εκθέσεις διαχωρίζονται. Τα μηνύματα των δύο εκθέσεων θα πρέπει να τα συγκεράσουμε. Πράγματι, όταν ε, βλέπουμε τόσο πυκνές ρυθμίσεις όπως έχουμε τώρα για τις επιγραμμικές υπηρεσίες στο online και για το, όλο το, όλη τη, μαζική τηλεόραση θα πρέπει να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε όλα αυτά. Οι γραμμικές υπηρεσίες εξακολουθούν να ακολουθούν τις παλιές συνταγές για τη διαμόρφωση του προγράμματος και τα άλλα δεν είναι τόσο δυσδυτικά στην αγορά. Παρ' όλα αυτά όμως, αν δούμε τη συμπεριφορά των νέων που ε, μπαίνουν στο διαδίκτυο, δεν θα πρέπει να μείνουμε... Μπορεί να μην είναι κλασική τηλεόραση, αλλά έχουν τη δυσδυτικότητα ενός μαζικού μέσου πλέον. Οπότε θα πρέπει να το δούμε και αυτό. Ε, και αυτό είναι το βασικό πολιτικό ζήτημα. Δεν έχουμε τελεσίδικη απάντηση ακόμα. Τώρα ψάχνουμε να δούμε πώς θα τα χειριστούμε όλα αυτά. Ω ένα βαθμό λοιπόν συμφωνώ ότι καταρχήν πρέπει να αξιολογήσουμε θετικά την οδηγία με βάση συγκεκριμένους στόχους που είχαμε διατυπώσει, αλλά βλέπουμε και σαφή προβλήματα τα οποία τα είπατε, δεν εφαρμόζεται παντού, τα κράτη-μέλη έχουν διαφορετική σχέση με την οδηγία, ε, έχουμε έτσι κι αλλιώ ε, συμφωνήσει μόνο σε ελάχιστα πρότυπα, αλλιώ δεν θα είχαμε συμφωνήσει, άλλα κράτη-μέλη τα ξεπερνούν αυτά, άλλωστε αυτό είχε προβλεφθεί. Ε, αυτό που είπε η Πέτρα Κάμερ Τέφερτ και ο κύριος Μπόρις, η ε, δύναμη που έχουν τα τετελεσμένα γεγονότα. Εμείς ε, μιλάμε για διαφημίσεις 12 λεπτών, πολλές φορές παρακάμπτεται. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι εποπτικοί φορείς, τα εποπτικά συμβούλια συμπεριφέρονται στο ρυθμιστικό τους ή παρεμβατικό τους ρόλο όπως θέλουμε και όπως έχουμε συμφωνήσει σε πολιτικό επίπεδο για τον πλουραλισμό των μέσων και αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ η συγκέντρωση των ΜΜΕ θα πρέπει να δούμε πολύ προσεκτικά στη φάση των διαβουλεύσεων τι στάση θα κρατήσουμε εδώ και πώς θα συνεργαστούμε και με άλλες επιτροπές όπως την ΛΥΜΠΕ. Ε, κάτι άλλο επίσης ε, που πρόσεξα. Αναφέρατε το παράδειγμα της Άξα στη Γαλλία και το αντισημιτικό περιεχόμενο και την Oitelzat που φρόντισε να μην διαδοθούν όλα αυτά. Αυτό το βρίσκω σωστό. Ξέρω ότι η Oitelzat σε σχέση με την Κίνα επίσης ακολούθησε συγκεκριμένη πολιτική που αφορούσε το δημοκρατικό περιεχόμενο και όχι τον αντισημιτισμό. Αυτό είναι λιγότερο ε, σωστό. Ε, για να μην πω ότι ήταν λάθος η πολιτική αυτή. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι ρυθμίσεις συζητάμε κάθε φορά και τι θέλουμε να προχωρήσουμε, να, να ε, προβάλλουμε σε ε, κοινωνικό επίπεδο. Αλλά παράλληλα το Ιράν ή την Κίνα ή αυταρχικά δικτατορικά καθεστώτα δεν θα πρέπει να τα ε, ενθαρρύνουμε. Και αυτό είναι ένα καθήκον της ρυθμιστικής μας πολιτικής, να ορίσουμε πολύ συγκεκριμένα τι θα πρέπει να καταδικάζουμε και τι όχι. Αυτά από τη δική μου την πλευρά. Για να δούμε τώρα, η κυρία Κώστα βλέπω ότι ζητεί το λόγο. Παρακαλώ να ευχαριστήσω θα ήθελα τον συνάδελφο Μπόρις, διότι νομίζω πως ε, έριξε άπλετο φως στη, στα σημεία της εκθέσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και να υπογραμμίσω τρία τεινά θα ήθελα. Μου φαίνεται ότι είναι σωστό αυτό που υπόθηκε ότι συνολικά η οδηγία με όλα της τα στοιχεία θα πρέπει μάλλον να απευθύνουμε έκκληση στα κρατη μέλη να εφαρμόσουν τις βασικές της πτυχές. Θα πρέπει όμως να εξυγχρονιστεί, να ενημερωθεί. Διότι υπάρχει και αυτό το πανόραμα το οποίο εξή περιγράψετε προηγουμένω και πολύ καλά μάλιστα. Αλλά να σε υπόψη την κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη, όπω και το δικό μου βεβαίω, διαπιστώνονται μεγάλε αμέλειε όσον αφορά την εφαρμογή τη. Πλουρασμό των μέσων καταρχήν. Εδώ αναφέρθηκε η ουγγρική περίπτωση στην έκθεση. Αλλά και η Ιταλική θα μπορούσε. Διότι νομίζω πω είναι ένα πολύ σημαντικό το ζήτημα αυτό. Κατά την έννοια ότι υπάρχουν κάποιε πτυχέ, Αναφέρομαι στο τράστο κάθετο, το οποίο δεν αξιολογείται. Την συγκέντρωση η οποία προκύπτει όχι μόνο, αλλά και από τη συγκέντρωση της διαφήμισης, από την οποία εξαρτάται και σε μεγάλο βαθμό ο πλουραλισμός στην τηλεόραση. Νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να εξειδικευτούν πολύ περισσότερο Τουλάχιστον ω προ το ερμηνευτικό, δεν λέω τροποποιώντα την οδηγία. Διότι βεβαίω κάτι που δεν λειτουργεί και δεν μπορεί να λειτουργήσει, αν πολύ δύσκολα μπορεί αν θέλετε να καλυφθεί και αυτό το θέμα. Δεύτερον, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή διότι όλοι μας γνωρίζουμε και πολύ καλά μάλιστα ότι οι τηλεοράσεις δεσμεύονται, είναι υποχρεωμένες να παράγουν και διανέμουν μια, ένα ποσόστοση ευρωπαϊκών προγραμμάτων, είτε εθνικών και μη εθνικών, και να επενδύσουν το 10% της δικής τους, ε, του δικού κύκλου στην ανεξάρτητη παραγωγή. Πρόκειται για περιπτώσεις δηλαδή όπου οι τηλεοράσεις, είτε οι εμπορικέ είτε οι κρατικές, όταν συμπαράγουν προγράμματα με ανεξάρτητες ανεξάρτητους παραγωγούς αποκτούν αυτά τα δικαιώματα για πάντα. Δηλαδή δεν υπάρχει μια δέσμευση, μια υποχρέωση η οποία δεν καθιστά εκχωρήσιμα όλα τα δικαιώματα. Επομένως, όταν πρέπει κατόπιν να γίνει η διανομή, η πώληση προϊόντων, τηλεοπτικών προϊόντων, η πρόσβαση Φερρυπίνες σε ευρωπαϊκά ε, προγράμματα, οι ανεξάρτητοι φορέ δεν έχουν δικαίωμα. Δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή μετάδοση και τι ευρωπαϊκέ συμπαραγωγέ. Πρόκειται συνεπώ για δεδομένα και στοιχεία, τα οποία φαντάζομαι δεν είναι οι αρχέ δηλαδή που λείπουν από την οδηγία αυτή, αλλά κάποιε διευκρινήσει που πρέπει να δοθούν. Και εύχομαι ότι και στο πλαίσιο τη δική μα νομοδοτήσεω, του συναδέλφου Μπόρι δηλαδή, θα μπορούσαμε να ζητήσουμε μια περαιτέρω διευκρίνηση. Και τρίτον, σε ό,τι αφορά τη διαφήμιση, δεν υπάρχει ούτε μια αφιβολία. Ότι λέγεται βεβαίω τώρα εδώ ότι όλα τα, στα καλό τα κράτη-μέλη διαπιστώνεται υπέρβαση των 12 λεπτών. Αλλά υπάρχει και αυτή η έμεση, υποβολημαία θα έλεγα μάλιστα, διαφήμιση που επιτρέπει να ξεπεραστεί αυτό το χρονικό όριο. Διότι δεν είναι διακρίσιμη και δεν είναι αναγνωρίσιμη αυτή η διαφήμιση ω τηλεοπτική διαφήμιση. Αναφέρθηκε και αναφέρεται η ισπανική περίπτωση. Και αυτό να πω κάτι θα ήθελα να μου επιτρέπετε, διότι υπάρχει και δεν ξέρω αν αυτό αναφέρει στην οδηγία, ίσως ο Μπόρις ε, να μου πει αν υπάρχει αυτή η ερμηνεία στην οδηγία αυτή. Αλλά μια κατάσταση, σε κατά που πάρα πολύ αρνητική και θα έπρεπε να επισημανθεί, είναι ότι ήδη οι πρωταγωνιστές των μεταδόσεων αυτών στον διαφημιστικό χώρο γίνονται διαφημιστική αν θέλετε χρηματοδότηση. θυμίζω ότι στην Ιταλική νομοθεσία αυτό απαγορεύεται. Αλλά αυτό βεβαίω είναι ένα φαινόμενο αρκετά διδεδομένο. Και θα ήθελα να ξέρω αν αυτό προβλέπεται ω πιθανό όριο κατά την ερμηνεία τη οδηγία αυτή. Και πολύ καλό είναι αυτό που γίνεται εδώ, η διάκριση, αν θέλετε, και που αναφέρω εδώ οι σαξιστικές, που είναι εικόνες στη τηλεόραση που πρέπει και οπωσδήποτε ε, να ελέγχονται και να καταπολεμηθούν και να καταπολεμούνται. Και νομίζω ότι θα πρέπει να προωθήσουμε και περαιτέρω αν θέλει κώδικες αλλά και να υπάρχει και ένα governance, μια διακυβέρνηση με... στην οποία θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των χρηστών που θα έχουν ευξημένο ρόλο έναντι των αρχών. Αλλά σε ό,τι αφορά τι ε, τηλεοπικοινωνικέ αρχέ καλό θα ήταν να τι ακούσουμε, διότι νομίζω πώ έχουν κάτι να μα πούν. Δηλαδή ότι οι αρχέ των διαφόρων χωρών που ασχολούνται δηλαδή και επιτηρούν με τι τηλεοπτικέ παραγωγές και τι εκπομπέ. Θα πρέπει νομίζω ο εισηγητή να δει αν θα έπρεπε να ακούσει την άποψή του ή αν σε αυτή την γνωμοδότηση, δεν ξέρω αν ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί νομίζω πραγματικά ότι είναι μια φωνή που πρέπει να γίνει ακουστή και να την ακούσουμε, διότι έχει σχέση με την εφαρμογή τη οδηγία και ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελε ο κύριος Μπόρις να παρέμβει, μετά θα παρέμβει η Επιτροπή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις τους, τα σχόλιά τους. Ε, ιδιαίτερος που οι δύο ε, διαφορετικές εκθέσεις που συντάσσουμε θα είναι συμβατές η μία με την άλλη, συνεκτικές, γιατί και οι δύο εξάλλου εστιάζονται στο προκλήσεις του μέλλοντος στον τομέα των κουστικών μέσων. Πρέπει βέβαια να δείξουμε υπευθυνότητα και να μην ανοίξουμε το δρόμο σε μια υπερβολική, υπερβολικά παρεμβατική πολιτική. Ας μην ξεχνάμε ότι ο ρόλος μας είναι να διασφαλίζουμε τα ελάχιστα πρότυπα προστασίας, αλλά πρέπει να παραμείνουμε και να δείξουμε υπευθυνότητα. Και έτσι ώστε ό,τι και αν προτείνουμε αυτό να μην δημιουργήσει αντιδράσεις, Συμφωνώ πάντως ότι πρέπει να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως για παράδειγμα αυτές που μας θέτει η υβριδική τηλεόραση ή αυτά που αναφέρατε εσείς σε σχέση με την επίβλεψη, την εποπτεία και την σχέση, το ρόλο μάλλον των εθνικών ε, ραδιοτηλεοπτικών συμβουλίων. Θα μπορούσαν αυτά τα συμβούλια στη συνεργασία και με την Επιτροπή να δημιουργήσουν κανόνες διοντολογίας, ε, κανόνες για το διαφημιστικό χρόνο, όρια, ε, κανόνες που να ρυθμίζουν ζητήματα σε σχέση με την μυσαλλοδοξία ή τα σεξιστικά μηνύματα. Η ε, βρήκα θετική ανταπόκριση την Επιτροπή και θεωρώ ότι πρέπει να συζητάμε αυτά τα ζητήματα ανοιχτά. Τώρα, όσον αφορά τον πλουραλισμό και την καταπολέμηση των μονοπωλίων, τα αντιμετωπίζω όλα αυτά τα θέματα στην ε, γνωμοδότησή μου και σας ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Θα τα λάβω υπόψη. Ευχαριστώ, κύριε Μπόρις. Τώρα θα ήθελα να ζητήσω από τους εκπροσώπους της Επιτροπής, η κυρία Αντεπτούα και ο κύριος Μασέλ. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και τον εισηγητή και τα μέλη του Κοινοβουλίου που δείχνουν τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη γνωμοδότηση που είναι ε, επί της πρώτης έκθεσης που παρουσιάζει η Επιτροπή στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Θα προσπαθήσω συνοπτικά να παρουσιάσω τις απόψεις μου για να μην επαναλάβω αυτά που ήδη υπόθηκαν, αλλά κυρίως να εστιάσω σε κάποια θέματα που θεωρώ σημαντικά και μπορούν να αποτελέσουν τροφή για συζήτηση. Όπως εξηγήσατε κι εσείς, η έκθεση αποτελείται από δύο μέρη που εξηγεί και τον λόγο που υπήρξε αυτή η καθυστέρηση στην υποβολή της. Χρειαζόταν η ε, περισσότερος χρόνος και περισσότερη έτσι, εργασία προκειμένου να ασχοληθούμε με τα ζητήματα των χρηστών. Το πρώτο μέρος λοιπόν κοιτά αναδρομικά πώς εφαρμόστηκε η οδηγία την περίοδο 2009-2011 και ένα δεύτερο μέρος της έκθεσης αφορά στο μέλλον πώς μπορούμε να καλύψουμε τα νέα μέσα και τις ε, νέες τεχνολογίες που αναπτύσσονται προς το πρώτο μέρος, το παρελθόν. Υπενθυμίζω ότι αυτή η οδηγία αφορά ζητήματα εσωτερικής αγοράς ρύθμιση την παροχή υπηρεσιών στην ενία αγορά και αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει να υπάρχουν σχεδόν 8.000 πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια αγορά σε πλήρη άνθηση και δεδομένων των ε, οικονομικών προβλημάτων είναι εντυπωσιακό το περιεχόμενο, το, το, το εύρος του περιεχομένου που προτείνεται. Εδώ υπάρχει και ζήτημα εναρμόνισης και ζήτημα επικουρικότητας, μια και πρόκειται για οδηγία ενίας αγοράς, αλλά επίσης και θέματα που άπτονται της προστασίας σημαντικών αξιών της κοινωνίας, Όπω αυτά που αναφέρατε και εσεί, η προστασία των ανηλίκων και η καταπολέμηση της μυσαλλοδοξία. Και σε αυτό το πλαίσιο η Επιτροπή λειτουργεί ως θεματοφύλακας των ε, συνθήκων, ιδιαίτερα στην περίπτωση του ε, Αλαξά αυτών των εκπομπών. Η Επιτροπή κινητοποιήθηκε με από την ε, παρέμβαση της Γαλλίας καθότι το ε, τηλεπτικό αυτό κανάλι του Αλαξά βρισκόταν ε, υπό την νομική δικαιοδοσία της Γαλλίας. Επίσης υπόκειτο και στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο επειδή το Sat είναι Ευρωπαϊκός Δορυφόρος και αξιοποιώντας αυτό το δίκαιο απαγορεύτηκαν αυτές οι εκπομπές. ο ορισμός του ποιο περιεχόμενο μπορεί να θεωρηθεί απαγορεύσιμο ή επιτρέψιμο δεν είναι κάτι που είναι εναρμονισμένο στο ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι, ε, ρυθμίζεται σε εθνικό επίπεδο. Και εδώ ε, επισέρχεται η αρχή της ε, επικουρικότητας σε αυτήν την οδηγία. Αλλά στην συγκεκριμένη περίπτωση του Αλαξά δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι έπρεπε αυτό το περιεχόμενο να απαγορευτεί. Είναι περιορισμένες οι δυνατότητες για εξαιρέσεις, για παρεκκλήσεις ε, σε αυτήν την οδηγία. Και το τελευταίο στοιχείο που αφορά στις διαφημίσεις, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, προσπαθεί η Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την διαφημιστικά μηνύματα παρακολουθούμε μια... Ε, ε, ε, έχουμε ένα δείγμα κρατών μελών που το ανανεώνουμε τακτικά προσπαθώντας να παρακολουθούμε επί δύο μήνες, 24 ώρες το 24ωρο περίπου 300 κανάλια, άρα μιλάμε για πολλά διαφημιστικά μηνύματα τα οποία αναλύουμε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της παρακολούθησης διαπιστώνουμε ορισμένες παραβιάσεις. Και διαπιστώνουμε επίσης και την εξέλιξη της διαφήμισης, νέες μορφές διαφήμισης που εμφανίζονται και που θέτουν ερωτήματα όσον αφορά την πρακτική των διαφημεζόμενων και την ποιότητα Ίσως λοιπόν θα χρειαστεί μια ε, ενημέρωση, μια επικαιροποίηση της ανακοίνωσης για την διαφήμιση για να δούμε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις νέες πρακτικές των, της διαφήμισης μένοντας πιστοί στο πνεύμα της οδηγίας. επίσης σε σχέση με την ε, διαφήμιση όσοι ενημέρωσης της Επιτροπής συμπεριλάμβανε και, και ένα ποιοτικό στοιχείο, μια αξιολόγηση ποιοτική της διαφήμισης και του κατά πόσον είναι επαρκής ε, το ρυθμιστικό πλαίσιο, επαρκές το ρυθμιστικό πλαίσιο. Θα βρείτε σχετικά στοιχεία στην έκθεσή μας. Υπάρχουν λίγες παραβιάσεις σε, στο επίπεδο της ποιότητας, αλλά ανάλογα με το κράτος μέλος βλέπουμε διαφορετικά στοιχεία της ε, οδηγίας να παραβιάζονται πιο συχνά, να εμφανίζονται πιο συχνά σε αυτά τα τύπου τα ερωτήματα. Και αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο, το οποίο θα το διερευνήσει περισσότερο η Επιτροπή. Μέχρι εδώ λοιπόν είχα να σας πω για το πρώτο μέρος της έκθεσης το που αφορά στην εφαρμογή της οδηγίας μέχρι το 2011. Δεν θα μπω στα, μεγάλη, μείζωνα σημασία ε, ζητήματα γιατί υπάρχουν και πιο αναλυτικές εκθέσεις. Ε, για παράδειγμα για την εφαρμογή των άρθρων 13, 16 και 17 Και έρχομαι τώρα στο μέλος, μέρος της έκθεσης που αφορά στο μέλλον. Βλέπουμε μάλλον μία σύγκληση. Εμφανίζονται νέες μορφές οπτικοακουστικών μέσων που δεν ε, καλύπτονταν από την οδηγία. Αυτά τα, αυτές οι νέες μορφές έρχονται στο καθιστικό μας και πρέπει να δούμε πώς θα ανταποκριθούμε και εμείς σε αυτές τις νέες υπηρεσίες. Η μικρή οθόνη, αν και καταρχήν εμφανίζεται ως πάροχος ενός συγκεκριμένου περιεχομένου, βλέπουμε και άλλες υπηρεσίες να συνδέονται με αυτήν. Σε αυτή τη στιγμή η Επιτροπή προσπαθεί να αξιολογήσει με τελείως ανοιχτό πνεύμα την κατάσταση. Το πρώτο μέρος, το, το πρώτο εξάμεινο του 2013 θα είμαστε σε θέση να εκδώσουμε ένα κείμενο πολιτικής επί αυτών των θεμάτων. Ευχαριστούμε την Επιτροπή. Επομένως, το προσχέδιο γνωμοδότησης θα είναι έτοιμο στις 8 Δεκεμβρίου και θα ψηφίσουμε 21 Φεβρουαρίου 2013. Επομένω, τότε θα μπορέσουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα στρατηγικά ζητήματα και προχωράμε στο επόμενο σημείο τη σημερινή διάταξη. Που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τους Ντάνιελ Βέρτεν, Ρενάτα Κοπίνοβα και την κυρία Ελευθερία Μακρύ που είναι οι τιμηθέντες με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για την νεολαία 2012. Ε, το τελευταίο σημείο λοιπόν στην ημερήσια διάταξή μας σήμερα είναι να ακούσουμε αυτούς τους νικητές του Ευρωπαϊκού Βραβείου Καρλομάγνου για την νεολαία. Σας υπενθυμίζω ότι αυτό το βραβείο θεσπίστηκε το 2008 σε συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με το ε, Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου απευθύνεται σε νέους μεταξύ 16 και 25 ετών με στόχο την προαγωγή της ευρωπαϊκής και διεθνούς κατανοητικής. Προωθεί ε, προγράμματα, εγχειρήματα που έχουν υλοποιηθεί από κοινού από Ευρωπαίους νέους σε πάνω από δύο κράτη μέλη. Η επιλογή των προγραμμάτων έγινε σε δύο στάδια, πρώτα σε εθνικό επίπεδο ε, αποτελούμενο από έναν, ένα μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο των φορέων νεολαίας των κρατών μελών. Θα σας καλωσορίζω, καλωσορίζω τους νικητές αυτού του βραβείου, τους τιμηθέντες με αυτό το βραβείο. Και θα ξεκινήσουμε με τον Ντάνιελ Βερτά, που ε, κέρδισε το, την τρίτη θέση από την Ουγγάρια. Ladies Κυρίες και κύριοι, θα σας παρουσιάσω το τρίτο βραβείο του Καρλομάγνου, μια σύντομη εισαγωγή για το Psych Home Home και μετά θα εξηγήσω την επιτυχία του προγράμματος που οδήγησε στο βραβείο και με τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι ένα ε, πρόγραμμα ε, ταινιών ντοκιουμαντέρ για έναν φοιτητή που αποφασίζει μετά το Εράσμους να γυρίσει με το ποδήλατο στο σπίτι του και πάει από τη Μαδρίτη στη Βουδαπέστη, γυρίζοντας πίσω. Υπολογίσαμε ότι θα ήταν 2.700 ε, τα χιλιόμετρα που θα διένυε, αλλά στο τέλος ε, έγιναν αυτά 3.284 χιλιόμετρα πήγε από την Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, ε, Σλοβενία και μετά έφτασε στην ε, πατρίδα του μετά από περίπου 87 μέρες. Και βέβαια γυρίσαμε πολύ φιλμ καθοδόν. Παρακολουθείτε λοιπόν ο Λεβί στην ταινία μέχρι το τέλος. Δύο μέλη είχε το επιτελείο, ο κινηματογραφιστής Μαρτέμπαλο και εγώ ως διευθυντής και παραγωγός της ταινία. Η ιδέα μας ήταν ε, χωρισμένη στα δύο, δύο βασικά σημεία. Θέλαμε να φτιάξουμε μία ταινία, αλλά πιο σημαντικό ήταν ότι θέλαμε να δημιουργήσουμε μία κοινότητα νέων ανθρώπων από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο για να τους δείξουμε ότι μπορούν τα πράγματα να γίνονται διαφορετικά αν φεύγουμε από τα, την πεπατημένη. Ήθελα να σας πω ότι δεν είναι περιβαλλοντικό το, πρόγραμμα, το έργο αυτό, αλλά θέτει και περιβαλλοντικά θέματα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θέλει να ε, προωθήσει λίγο τη νέα δική μου γενιά που δεν είναι καθόλου τεμπέλικη. Η επιτυχία δείχνει ότι μπορούμε να κινητοποιηθούμε. Ε, δεν ε, ε, τα κάνουμε όλα αυτά αποσκοπώντας κάπου, αλλά για να χαρούμε. Αυτό είναι σημαντικό. Δεν βλέπουμε μεγάλα πράγματα, δεν ε, είμαστε κινηματικοί. Γράφουμε απλώ και δουλεύουμε για, να, για την αναψυχή μας. Όμως μπορούμε έτσι να ε, κινητοποιήσουμε πολλούς. Η απήχηση μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα ήταν σε πάνω από 150.000 ανθρώπους. Είχαμε screening σε πολλές χώρες, την Ολλανδία, τη Γαλλία, την ε, Ρωσία, τη Βραζιλία, την Ουγγαρία βεβαίως ε, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και τώρα περιμένουμε και πολλά φεστιβάλ να ανταποκριθούν ε, μετά από τις διακρίσεις που πήραμε. Θέλω να σας πω επίσης ότι εφαρμόσαμε νέο τρόπο κινηματογραφίας που είναι πολύ ενδιαφέρον θεωρώ γιατί συμμετείχε το ακροατήριο σε όλη τη διαδικασία. Συνήθως μέχρι τώρα όταν γυρίζουμε ένα φιλμ κατά τα γυρίσματα δηλαδή δεν μπορούσαν να συμμετέχουν οι παρευρισκόμενοι και το ακροατήριο αλλά τώρα με τα κοινωνικά μέσα αυτό γίνεται πια κάθε μέρα ε, είχαμε βίντεο για να ξέρει και η κοινότητα τι γίνεται και μπορούσαν να συζητήσουν όλο το εγχείρημα μαζί μας. Και έτσι μια ολόκληρη κοινότητα ε, κινητοποιήθηκε να χρησιμοποιεί ποδήλατο και πολλοί από αυτούς που συναντήσαμε στα κοινωνικά δίκτυα ε, ενθουσιάστηκαν και βγήκαν και εκείνοι με το ποδήλατο. Θέλουμε στο μέλλον να οικοδομήσουμε ακόμα περισσότερο αυτή την κοινότητα γιατί νιώθουμε υπεύθυνοι για αυτά που φτιάξαμε. Το βραβείο Καρλομάγνου ήταν μεγάλη βοήθεια γιατί το έργο είναι αυτοχρηματοδοτούμενο 100% και χωρίς την ηθική και οικονομική υποστήριξη του Ιδρύματος ε, δεν θα ήταν δυνατόν να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω όλους και αν έχετε ερωτήσεις Ευχαρίστως να τις απαντήσω. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτό ήταν το τρίτο βραβείο, το οποίο έλαβε 2.000 ευρώ ως βραβείο. Θα ακούσουμε τις τρεις παρουσιάσεις πρώτα και μετά να κάνουμε ερωτήσεις ή να κάνουμε σχόλια. Πάμε στο δεύτερο βραβείο, 3.000 ευρώ. Η Ευρώπη χρειάζεται σχολεία. Έχετε το λόγο. Η ε, Ρενάτε, Ρενάτα Κοπρίκοβα. Ε, λέγομαι Ρενάτα Κοπρίκοβα και θέλω να σας παρουσιάσω το έργο μας, ε, το οποίο είναι η ε, Ευρώπη κάνει σχολείο, φτιάχνει σχολείο στην Πράγα. Λέγεται Ευρώπα Ντέλα Σκόλου, Πράγα. Θα ξαναρχίσω. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, λέγομαι Ρενάτα Κοπρίβοβα και θα σας παρουσιάσω το πρόγραμμα Ευρώπα Ντέλα Σκολού, Πράγα, η Ευρώπη φτιάχνει σχολεία στην Πράγα. Το πρόγραμμα αυτό, από, ήδη από το 2008, επιτρέπει στους φοιτητές του προγράμματος Εράσμου ε, στο Πανεπιστήμιο του Καρόλου στην Πράγα να ε, συναντήσει παιδιά σε τσεχικά σχολεία και να μάθει περισσότερα για το σύστημα εκπαίδευσης και το σχολικό σύστημα στην Τσεχία, ενώ προετοιμάζουν εθελοντικά προγράμματα για τα μαθήματα, παρουσιάζοντας τον εμπολιτισμό της χώρας τους. Οι φοιτητές Εράσμου πολλές φορές ε, είναι απομονωμένοι μεταξύ τους. Έτσι όμως έχουν τη δυνατότητα στη χώρα που θα πάνε για ένα ή δύο εξάμηνα να μάθουν πολλά πράγματα και να δείξουν και στα παιδιά τον πολιτισμό της δικής τους χώρας με τη σειρά τους. Η ιδέα για αυτό το πρόγραμμα προέρχεται από τον εταίρο μας, ε, το Γερμανικό Σύλλογο «Η Ευρώπη φτιάχνει σχολείο», με το οποίο τη συγκατάθεση εμείς χρησιμοποιήσαμε την τσεχική μετάφραση το, από τα γερμανικά για το όνομά μας, δηλαδή κάναμε το Ευρώπα Αντέλα Σκόλου. Αυτό που μας διαφοροποιεί είναι ότι τα προγράμματα κατά μέσον όρο ε, διαρκούν τρεις ε, ώρες διδασκαλίας και τα περισσότερα ε, μεταφράζονται από το, την αρχική γλώσσα στα τσεχικά από φοιτητές τσέχους ε, που έχουν επίτιμη δραστηριότητα. Για την οργανωτική πλευρά ε, ασχολείται το, η ομάδα Εράσμους στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πράγας που ενημερώνει πάντα τους φοιτητές του Εράσμου με email για τη δυνατότητα να προετοιμάσουν κάποια τέτοια προγράμματα και εκείνοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται ε, παρουσιάζονται με τα, τις θεματικές τους προτάσεις, τις υποβάλλουν σε εμά και μετά οι θεματικές προτάσεις στέλνονται στα σχολεία που συνεργάζονται και επιλέγονται τα θέματα αν ταιριάζουν στο μάθημα καλά ή αν πιστεύουν ότι θα είναι ενδιαφέροντα τα θέματα για τους ε, μαθητές. Ο φοιτητή του Εράσμου κατά κανόνα συνοδεύεται από έναν φοιτητή Τσέχο που ε, κάνει τη διερμηνία άμα δεν καταλαβαίνουν οι μαθητές. Καμιά φορά οι φοιτητέ ε, προετοιμάζουν από κοινού τα προγράμματα με τους επόπτες του Τσέχους, αλλά αυτό εξαρτάται από το πρόγραμμα. Ε, τώρα σε εμά, στην ομάδα Εράσμου, υπάρχουν περίπου 15 Τσέχοι φοιτητέ που διερμηνεύουν ε, τακτικά για τα προγράμματα και ελπίζουμε ότι ο αριθμός του συνεχώς θα αυξάνεται. Τώρα, σε ποια γλώσσα θα τρέξει το πρόγραμμα αυτό εξαρτάται από τη συνεννόηση που θα γίνει με το σχολείο. Αν είναι η μητρική γλώσσα του φοιτητή Εράσμου ε, μία γλώσσα που διδάσκεται στο σχολείο, τότε θα γίνει σε αυτή τη γλώσσα. Αν όμω μιλάει ο φοιτητή Εράσμου ελληνικά, φιλανδικά ή ουγγρικά, τότε γίνονται τα προγράμματα κατά κανόνα στα αγγλικά. Ω ε, σχολές συνεργαζόμενε, σχολεία δηλαδή, έχουμε περίπου 15, αλλά ε, κάνουμε προσπάθεια να αυξήσουμε τον αριθμό, ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε. Τα περισσότερα συνεργαζόμενα σχολεία βρίσκονται στην Πράγα, αλλά και σε μικρότερες πόλεις κοντά στην Πράγα, στο Βάλσιμ, στο Μπένεσοφ, στο Ρίκα, Ρίτσανη. Ε, οπότε κάνουν και μια μικρή εκδρομή για να φτάσουν εκεί. Χαιρόμαστε γιατί αυτό το πρόγραμμα ε, συγκεντρώνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Το, αρχίσαμε το 2008-2009 και είχαμε μόνο τέσσερα προγράμματα. Το 2010-2011 είχαμε 29 και πέρσι το 2011-2012 είχαμε 36 και τώρα, μέχρι τώρα έχουμε υποπροετοιμασία 30 προγράμματα τα θέματα των ε, προγραμμάτων ε, είναι σε σχέση με τον πολιτισμό, την τέχνη, την ιστορία, λογοτεχνία. Ε, ο γερμανικός εξυπρεσιονισμός ήταν ένα από αυτά τα προγράμματα, ή προσωπικότητες από την Πολωνία, η Ιταλική τέχνη. Κάποια ενδεικτικά σας αναφέρω. Τα προγράμματα κατά κανόνα ολοκληρώνονται είτε με μια αφίσα, ένα πλακάτι ή με προετοιμασία ενός μικρού θεατρικού έργου, το οποίο και παρουσιάζεται στο σχολείο Τέλος θα ήθελα να σας πω ότι χαιρόμαστε διότι με αυτή την εθελοντική δραστηριότητα καταφέραμε να καταδείξουμε τις διαφορές και τις ομοιότητες μεταξύ ημών Ευρωπαίων που αποτελούν την ευρωπαϊκή κοινή μας κληρονομιά τα αναδείξαμε όλα αυτά και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τον κοινό διάλογο. Η δεύτερη θέση στο βραβείο Καρόλου για τους νέους μας βοήθησε να δείξουμε το πρόγραμμα αυτό. Η Ευρώπη φτιάχνει σχολείο όχι μόνο στην Τσεχία αλλά σε όλη την Ευρώπη και θα χαιρόμαστε αν ενδιαφερθούν για την ιδέα αυτή οι άνθρωποι και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Θα ήταν πραγματικά καταπληκτικό αν από αυτή την απλή ιδέα προέκυπτε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ.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 Ε, I come from Athens. My name is Elena Makri and I'm a journalist. Ε, I bet you, you come... Είμαι από την Αθήνα, είμαι δημοσιογράφος. Είμαι σίγουρος ότι έρχεστε πολύ συχνά σε επαφή με, τις, με δημοσιογράφους, αλλά σήμερα θα σας μιλήσω για ένα καινοτόμο πρόγραμμα ε, δημοσιογραφίας από νέους. Ε, είναι κάτι που δεν το κάνουμε συχνά στον τομέα του τύπου να έχουμε καινοτομίες στην Ευρώπη είτε μας αρέσει είτε όχι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης διαμορφώνουν την άποψή μας για τον κόσμο, διαμορφώνουν την αντίληψή μας για τα πράγματα. Γι' αυτόν τον ε, λόγο θεωρούμε ότι η δημοσιογραφία, η διερευνητική δημοσιογραφία πρέπει να είναι υπέρ του, λειτουργεί υπέρ του δημόσιου συμφέροντος. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ο τρόπος με τον οποίο καλύπτεται δημοσιογραφικά σε παγκόσμιο επίπεδο η οικονομική ε, κρίση. Έχουμε άρθρα τα οποία αλληλοκατηγορούν, ε, κατηγορούν μάλλον οι Έλληνες τους Γερμανούς, τους, τους ονομάζουν Ναζί και αντιστρόφως οι Γερμανοί κατηγορούν τους Έλληνες ότι είναι τεμπέληδες. Συνέχεια έχουμε δημοσιεύματα που αναφέρονται στην πιθανότητα να εγκαταλείψει την Ευρωζώνη ένα κράτο Όλα αυτά είναι προπαγάνδα, οδηγούν σε εύκολα και απλοϊκά συμπεράσματα, ισοποδώνοντας την πραγματική πολυπλοκότητα του προβλήματος. Ποιος κερδίζει από αυτό το αυτή την κατάσταση, αυτή την, το μπέρδεμα, σίγουρα όχι η Ευρώπη. Πρέπει να το αλλάξουμε αυτό και θέλουμε στην Ευρώπη οι άνθρωποι να γνωρίζουν πολύ περισσότερο ο ένας για τον άλλον. Τι κάνουμε λοιπόν γι' αυτό. Δημιουργούμε δημοσιογραφικό περιεχόμενο που λειτουργεί υπέρ του δημοσίου συμφέροντος στην Ευρώπη. Στέλνουμε ε, φωτογράφους, ε, κάμεραμαν και δημοσιογράφους ε, σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Ο στόχος μας είναι εκεί οι άνθρωποι αυτοί να έρθουν σε επαφή άμεση με την τοπική κοινωνία, να δουν με ποιον τρόπο ζει ο κόσμος εκεί. Οι νέοι αυτοί ε, δημοσιογράφοι έρχονται στη θέση των άλλων Ευρωπαίων πολιτών, των άλλων Ευρωπαίων νέων. Αυτού του τύπου δημοσιογραφία κινδυνεύει γιατί όλο και περισσότερο θεωρείται πολυτέλεια. Έχουμε όλο και λιγότερους πόρους να διαθέσουμε στους δημοσιογράφους που θέλουν να διερευνήσουν σε βάθος τα ζητήματα. Συχνά έχουν να αντιμετωπίσουν ε, προβλήματα χρόνου και ας σας δώσω ένα παράδειγμα. Έχουμε έναν, τον Ευρωπαίο ανταποκριτή, τον ανταποκριτή ο οποίος βρίσκεται σε κάποια ευρωπαϊκή πόλη, στις Βρυξέλλες ας πούμε, και πρέπει να αντιμετωπίσει όλη την πραγματικότητα των ε, κρατών μελών της Μεσογείου. Αλλά η κατάσταση στις Βρυξέλλες είναι πολύ διαφορετική από την κατάσταση στις μεσογειακές χώρες. Έτσι υπάρχει ένα κενό, ένα κενό στο, στην κατανόηση, στην αντίληψη. Οι δημοσιογράφοι δεν έρχονται σε επαφή, δεν θέλουν να αναμειχθούν και πολύ με την τοπική κοινωνία. Εμείς λοιπόν αποφασίσαμε να αντιστρέψουμε τα πράγματα, να σκεφτούμε διαφορετικά είπαμε θα ε, ακολουθήσουμε μια άλλη μέθοδο που στα ελληνικά ονομάζεται μέθεξη. δηλαδή την ε, εσωτερική ε, επικοινωνία και την εσωτερήκευση της ταυτότητας του άλλου. Θεωρούμε ότι έτσι μπορούμε να προσφέρουμε πολύ περισσότερα και πολύ καλύτερες υπηρεσίες από τα δελτία τύπου, από τα τηλεγραφήματα του Reuters, του Associated Press κτλ. Αλλά ποια είναι η προστιθέμενη αξία για τους, για τους πολίτες από αυτά. Αυτό που προσπαθούμε εμείς να κάνουμε είναι να φωτίσουμε τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των Ευρωπαίων. Το δημοσιοποιούμε αυτά τα άρθρα σε μια ιστοσελίδα, το cafebubble.com. Θα σας δώσω και κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες. Αυτό που γίνεται είναι ότι στέλνουμε πάνω από 50 δημοσιογράφους σε 10 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες κάθε χρόνο. Προσπαθούμε να έρθουμε σε επικοινωνία και σε επαφή με τους ηγέτες της κοινωνίας των πολιτών. Αναφερόμαστε σε ζητήματα πολιτικής, κοινωνικά, οικονομικά και τρόπου ζωής και με αυτό τον τρόπο οι δημοσιογράφοι μας έχουν μια σημαντική δημοσιογραφική εμπειρία και μια σημαντική ευρωπαϊκή εμπειρία επιτόπου. Έτσι η Ευρώπη γίνεται πιο απτή ιδέα, πιο απτή για να την κατανοήσουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και θεωρούμε ότι έτσι συμβάλλουμε και στην αλληλοκατανόηση των Ευρωπαίων πολιτών. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσοι βοήθησαν στο εγχείρημα. Θέλω να σας ευχαριστήσω για το βραβείο. Αυτά τα χρήματα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμα και θέλω να ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό ε, Κοινοβούλιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει αυτού του είδους τη δημοσιογραφία. Thank you very much. And Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να συγχαρώ και προσωπικά και εξ ονόματος όλων και τους τρεις βραβευθέντες για το βραβείο αυτό του Καρλομάγλου για τους νέους. Είχα τη χαρά και την τομή κάποια στιγμή να είμαι στην ε, Γερμανική Επιτροπή για το βραβείο και πραγματικά ενθουσιάστηκα βλέποντας πόσα καταπληκτικά projects ε, αναδύθηκαν από κάτω και πόσοι ε, πολλοί νέοι Ευρωπαίοι σκέφτονται και προβληματίζονται πώς να φέρουν πιο κοντά την Ευρώπη με διάφορα ε, έργα, με θεατρικά, με ποδηλασίες, με προγράμματα για δημοσιογράφους. Υπάρχουν τόσα πολλά και διαφορετικά μέσα και τρόποι. θέλω να πω σε όλους τους βραβευθέντες ότι τα προγράμματα συνεχίζονται, πολλά από αυτά ε, είναι βιώσιμα και συμβάλλουν σε αυτό που θέλουμε όλοι, την ευρωπαϊκή συνείδηση, που δεν μπορούμε να την επιβάλλουμε και να την υπαγορεύουμε από τα πάνω, είναι κάτι που πρέπει να δημιουργηθεί από κάτω, από τη βάση. Αυτά τα προγράμματα εξυπηρετούν ακριβώς αυτό το σκοπό. Και είναι πάρα πολύ ωραίο ότι ασχολούνται οι νέοι και σκέφτονται τι ιδέες μπορεί να κατεβάσουν για να γνωριστούν αμοιβαία, να αναδείξουν διαφορές και ομοιότητες, πρώτα να τις δουν, να τις κατανοήσουν, να τις αποδεχτούν ότι υπάρχουν διαφορές, ότι υπάρχει μια ενότητα στην εταιρότητα. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι ε, θαυμάσιο που μπορούμε να το βλέπουμε ότι υπάρχει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ για τον ενθουσιασμό σας και εύχομαι να συνεχίσουν κι άλλοι στα βήματα τα δικά σας και να νιώσουν ότι θα εμπνεύσε, θα εμπνευστούν και άλλοι να ακολουθήσουν και να σας μιμηθούν. Έτσι, παρά τις δυσκολίες, παρά τις κρίσεις, ε, στο τέλος η Ευρώπη ε, θα τα καταφέρει. Ευχαριστώ, Πέτρα. Ο Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ως ε, εκπρόσωπος των ε, φιλελευθέρων δημοκρατών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους νέους για τις παρουσιάσεις τους, για τα project τους, τα έργα τους. Όπως επίσης και για την, ε, την ενεργό τους συμμετοχή. Ξέρουμε πως φτάσαμε στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα, ως Ευρώπη, αλλά το ερώτημα που τίθεται είναι ποια θα είναι τα, τα επόμενα μας βήματα. Και το ερώτημα αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολο. Γιατί αν δείτε νέους σαν για αυτούς και τα έργα τα οποία έχουν και, τα, ε, και τις ιδέες τις οποίες έχουν, για έναν ευρωβουλευτή όπως εγώ, μου δίνουν αισιοδοξία. Αισιοδοξία για το μέλλον. Όπως επίσης και μου προσφέρουν και μια ιδέα ότι έχουμε δηλαδή τις αξίες μας εμείς στην Ευρώπη, τις οποίες οι νέοι της Ευρώπης θα προσπαθήσουν να τις προωθήσουν και να τις ε, υπερασπιστούν και στο μέλλον. Γι' αυτό λοιπόν να σα ευχηθώ κουράγιο, κάθε επιτυχία στον δρόμο τον οποίο διαλέξατε να ακολουθήσετε και ελπίζω πραγματικά ότι θα συνεχίσετε να εργάζεστε για αυτόν τον πολύ καλό σκοπό διότι πραγματικά αποτελεί μια πρόκληση για όλους. Πρέπει να δούμε και να βρούμε τρόπους πώς θα ενισχύσουμε project τα δικά σας. Πώς μπορούμε να τα βελτιώσουμε για να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη του Ευρωπαίου πολίτη στο μέλλον του. Όπως επίσης και για να μπορεί να έχει έτσι μια πιο αισιόδοξη προοπτική για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ σε όλους σας και πάλι. Η κυρία Παλιαντέλη η κατόπιν κύριο Μπόλς. Το ελληνικά για να τιμήσω την Ελληνίδα που πήρε το πρώτο βραβείο, αλλά να συγχωράω το σύνολο των ε, βραβευτέντων για αυτή την ανική θετική ατμόσφαιρα που μεταφέρουν σε μια επιτροπή που πολεμάει για τους νέους, φροντίζει όσο μπορεί να ε, μειώσει τις επιπτώσεις που, έχουν, ε, που έχει στην καθημερινότητά τους η οικονομική κρίση στην Ευρώπη και που αγωνίζεται, ελπίζουμε να τα καταφέρει, να μην μειωθεί το ποσό που διατίθεται κάθε χρόνο για την ανταλλαγή ε, για το Εράσμους και ειδικότερα για την ανταλλαγή των φοιτητών που προέκυψε τις τελευταίες μέρες. Ε, το πιο σημαντικό για, τις, ε, για τη βράβευσή σας είναι ότι ε, μας βοηθάτε, ή μάλλον όχι, βοηθάτε τον Ευρω... τους ευρωπαϊκούς λαούς να δούνε διαφορετικά αυτή την πολυπολιτισμική συνύπαρξη και εκφράζοντας το μέλλον αυτής της προσπάθειας για μια ακόμη πιο ενωμένη Ευρώπη παρε... μας δίνεται μια αισιοδοξία που συχνά μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να επιστρέψω στην πρώτη βεβαιωτήσα ε, επηρεάζουν δραματικά και εμείς στην Ελλάδα το έχουμε βιώσει την ε, κατάσταση, κόβουν την αισιοδοξία, κόβουν την αγωνιστικότητα, μετατρέπουν ε, ζητήματα αυτογνωσίας σε, ε, πώς να πω, σε πολύ εύκολες διατυπώσεις του τι για όλα αυτά είναι οι άλλοι. Εμείς το βιώνουμε ε, στην Ελλάδα τα τελευταία τρία χρόνια. Πιστεύω λοιπόν ότι συμβάλλετε αποφασιστικά με τις προσπάθειές σας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το καταλαβαίνει. Ελπίζουμε ότι θα πληθύνουν αυτές οι προσπάθειες και ότι η προσπάθεια που γίνεται εδώ σε εμά μπορεί να πιάσει τους νέους ε, μέσα από εσά. Ευχαριστώ πολύ για όλους σας. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για τις παρουσιάσεις σας και τις θαυμάσιες ιδέες, διότι νομίζω πως η δημιουργικότητα και η φαντασία έχει μεγάλη σημασία. Και η αισιοδοξία δεν ήταν το μόνο στοιχείο που φάνηκε από τις παρουσιάσεις σας, διότι γύρω από τις ιδέες σας αυτές προσπαθήσατε, νομίζω, να προσελκύσετε όσο γίνεται και να ελκύσετε μάλλον όσο γίνεται περισσότερη προσοχή. Να φέρετε το πρόγραμμα έρασμου δηλαδή στο κατώτερο επίπεδο, στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορεί να φτάσει, στα σχολεία δηλαδή. Για να μπορέσουν κατόπιν και οι μαθητές να καταλάβουν τη σημασία, να εξοικειωθούν δηλαδή με νέους πολιτισμούς, να μάθουν νέες γλώσσες και μόλις τα εγκωδικεύσει και τα βάλετε αυτά τα μηνύματα στο μυαλό των νέων, θα παραμείνουν μαζί τους νομίζω για μεγάλο χρονικό διάστημα. Νομίζω πως αυτές οι ιδέες πραγματικά πρέπει να τύχουν της υποστήριξής μας. Και αυτό που είναι και το πιο σημαντικό είναι νομίζω η αισιοδοξία της νέας γενιάς. Διότι σήμερα ε, αποτινάσουμε όλα τα στερεότυπα. Όλα τα στερεότυπα που υπήρχαν και υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη γιατί νομίζω ότι αυτό αποτελεί ένα σημάδι των καιρών και πρέπει η νέα γενιά να αυτοοργανωθεί. Για μια ακόμη φορά λοιπόν ένα μεγάλο ευχαριστώ και σας εύχομαι συγχαρητήρια εκ βάθους καρδίας και ό,τι το καλύτερο για το μέλλον. Σας εύχομαι. So, um, the young winners, uh, you see... Οι νέοι λοιπόν νικητές. Είδατε πόσοι συνάδελφοι ικανοποιήθηκαν και πόσο ικανοποιημένοι είναι από τα δικά σας τα project. Ευχαριστώ πολύ λοιπόν και στα ελληνικά. Ελπίζω ότι θα παραμείνετε σε επαφή, γιατί είναι πολύ σημαντικό και για μα να ερχόμαστε σε επικοινωνία μαζί σα, με εσά του νέου δηλαδή, για να μπορέσουμε και να πείσουμε του συναδέλφου μα και του ανθρώπου δηλαδή, στο Συμβούλιο ότι σε κάποιο βαθμό χρειάζεται να γίνει περισσότερη δουλειά, όπω και εσεί δηλαδή, πράγμα το οποίο θα διευκολύνει και τι περαιτέρω εξελίξει. Φτάνουμε τώρα και επανερχόμαστε στο τελευταίο σημείο τη μεσαία διατάξεώ μα. το σημείο 10, έγκριση των αποφάσεων των συντονιστών. Οι συντονιστέ χθε το βράδυ πήραν κάποιες αποφάσεις οι οποίες στάλησαν εν συνεχεία με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Εγκρίνεται. Δεν νομίζω να υπάρχουν αντιρρήσεις. Η κυρία Παλιαδέλη, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μερικέ ερωτήσεις που αφορούν ε, στις αποφάσεις τις χθεσινές της, ε, των συντονιστών. Τις σέβομαι απολύτω και ξέρω ότι προκύπτουν μετά από απολύτω δημοκρατικέ διαδικασίε. Δεν τι αμφισβητώ επομένω. Θα ήθελα όμω να γνωρίζω και περιμένω να έχω την απάντηση από τους εκπροσώπους τους. Πρώτον, γιατί απορρίψαμε την... Είναι τρία ερωτήματα. Το πρώτο αφορά στην νομοθετική γνωμοδότηση για την... να το πω ε, στα, αγγλικά, όχι στα ελληνικά, για την τροποποίηση της απόφασης ΤΑΔΕ, της απόφασης ΤΑΔΕ και της απόφασης ΔΙΝΑ του Συμβουλίου με σκοπό την αύξηση του ποσοστού χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφυγών και ούτω ή άλλω. Και, και, και, λοιπά και λοιπά. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που ε, η Επιτροπή οριζόμαστε ως δικαιούχοι να καταθέσουμε μία γνωμοδότηση, γιατί την αρνιόμαστε. Θα ήθελα να γνωρίζω δηλαδή ε, ε για ποιο λόγο την απορρίψαμε, ενώ θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συμμετάσχουμε. Δεν ζητάμε εμεί να μπούμε σε έναν χώρο που δεν μα αφορά. Είναι ένα χώρο για τον οποίο ενδεχομένω μπορούμε να προτείνουμε μερικά, με μερικά επιχειρήματα πράγματα που ίσω συμβάλλουν σε αυτήν την θετική ε, ε, κίνηση του, να, μετά, να μετέχουμε σε αυτή την ε, γνωμοδότηση, μια τέτοια γνωμοδότηση. Θα ήθελα λοιπόν να ξανασκεφτούμε το ενδεχόμενο να ε, να κάνουμε τελικά τη γνωμοδότηση και προτείνω να την αναλάβω αν θέλετε. Ένα είναι αυτό το ερώτημα. Το δεύτερο είναι παρόμοιο. Στις ε, non-legislative reports ε, υπάρχει ένα, μία δυνατότητα να, να καταθέσουμε ως υπεύθυνη επιτροπή μία αναφορά σε σχέση με την ε, ενδιάμεση αξιολόγηση του Erasmus Mundus 2, ε, προγράμματος δηλαδή 2009-2013. Και εδώ καταλαβαίνω, παρόλο που είμαστε καθήλυνα αρμόδιοι, για ποιο λόγο δεν, ε, ε, δεν θέλουμε να κάνουμε μια τέτοια αναφορά. Και μια τρίτη ερώτηση, που είναι λίγο πιο ειδική, ε, επειδή στα πρακτικά δεν φαίνεται ο λόγος για τον οποίο, οι λόγοι για τους οποίους από τις προτάσεις για τις ε, αποστολές προτείνονται ορισμένες, ορισμένες πόλεις και απορρίπτονται μερικές άλλες θα ήθελα να γνωρίσω τον λόγο για τον οποίο αποκλείστηκε η Θεσσαλονίκη ε, όχι επειδή είναι η πόλη από την οποία προέρχομαι ή επειδή είναι ελληνική πόλη αλλά ως κατεξοχήν πολιτική ε, επιλογή. Θεωρώ ότι η, η περίοδος που περνούμε στην Θεσσαλονίκη θα ε, όφιλε να αντιμετωπιστεί από τους συντονιστές με μεγαλύτερη ενδεχομένως ευαισθησία σε ό,τι αφορά το timing. Ότι ίσως πρέπει να, κάτι που το βλέπουμε με τη σημερινή επίσκεψη της Μέρκελ στην, ε, της καγκελαρίου Μέρκελ στην Αθήνα. Σε τελευ... Δεν κρίνω τις αποφάσεις, θα ήθελα διευκρινήσεις για τον τρόπο με τον οποίο σκέφτηκαν οι συντονιστές, για να καταλήξουν σε αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ πολύ. Yes, Mrs. I, um... Κύριε Παλιαδέλη, με τα χαράς να απαντήσω στο ερώτημά σας και στις παρατηρήσεις σας. Οι συντονιστές είχαν λόγο για τις αποφάσεις τους. Να σας πω τον πρώτο, σε ό,τι αφορά το Ταμείο για τους Πρόσφυγες. Ο πολιτισμός ενδιαφέρεται ιδιαίτερα στην μετανάστευση, διότι η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει τους μετανάστες και να ενισχύσει επίσης και το πολιτιστικό διάλογο αλλά μιλούμε για ζήτημα, θέλετε, που έχει σχέση με την χρηματοδότηση από τον προλογισμό των προγραμμάτων για τους μετανάστες. Γι' αυτό το λόγο, λοιπόν, θα πρέπει να το αφήσουμε στην ΛΥΜΠΕ και στην, ε, στην ομάδα του προπολογισμού. Και επειδή είμαι εισηγήτρια εγώ στην Επιτροπή του Προπολογισμού, ξέρω ότι θα εργαστούμε πάνω σε αυτό το θέμα. Γι' αυτό το λόγο η Επιτροπή Πολιτισμού δεν θα πρέπει να ασχοληθεί αυτό. Θα πρέπει να γίνει σωστά ο επιμερισμό έργου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό είναι το επιχείρημα για την απόφαση την οποία λάβαμε χθε. Μου επιτρέψετε να, έχω την, να δηλώσω, να καταγραφεί η αντίρρησή μου, αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα, επομένω δεν το συζητάω. Ε, για τις άλλες δύο ερωτήσεις. Yes. On uh, the second point... Όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση για το ζήτημα σχετικό με το πρόγραμμα Erasmus, Πρόκειται για μια έκθεση όσον αφορά το πρώτο ίμιση της δεύτερης φάσης του Erasmus Mundus προγράμματος. Το Erasmus Mundus θα απορροφηθεί από το νέο πολιετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση και τον αθλητισμό των νέων. Τα μαθήματα που διδαχθήκαμε από το Erasmus Mundus θα ληφθούν υπόψη στην νομοθετική και την νομοπαρασκευαστική διαδικασία που θα δημιουργήσει και θα θεσπίσει το νέο πρόγραμμα. Και επειδή ακριβώ υπάρχουμε η μόνιμο εισηγήτη, η μόνιμη εισηγήτρια, οι συντονιστέ πήραν την απόφαση που έλαβαν χθε. Τελευταία ερώτηση, γενικής φύσεως, διότι είναι δουλειά των συντονιστών να παρουσιάσουν αυτό το οποίο επιθυμούν οι ομάδες. Και οι ομάδες παρουσιάζουν τα πράγματα όπως τα παρουσιάσαν χθε. Και σε ό,τι αφορά το ζήτημα το ποια είναι τα επόμενα μας βήματα, νομίζω ότι θα πρέπει να επισκεφτούμε τις δύο πολιτιστικές πρωτεύουσες ως συνήθως, γιατί συνήθως αυτό κάνουμε, για να ξέρουμε τι γίνεται εκεί. Στι δύο πολιτιστικέ πρωτεύουσε και κατόπιν ετέθηκε το ζήτημα ότι θα έπρεπε να εστιάσουμε την προσοχή μα και να εστιαστούμε σε χώρε και σε καταστάσει πρωτόγνωρε, που δεν έχουμε επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Και κατέστησε σαφέ ότι οι συγκεκριμένε αυτέ οι δύο προτάσεις που κάναμε λόγω πολιτιστικής ε, διαφορετικότητας στο βόρειο της Φιλανδίας είχαν τη σημασία τους και δεύτερον ήταν μια πολιτική χειρονομία για την Κροατία, γιατί τώρα προσχωρεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα έπρεπε να επισκεφτούμε την Κροατία. Δεν είναι ότι διαφορούμε και ότι δεν μας ενδιαφέρουν δηλαδή οι άλλες πολιτιστικές πρωτεύουσες και άλλες πόλεις οι ευρωπαϊκές. Είναι ότι πάμε σε ωραία μέρη και θέλουμε να πηγαίνουμε σε ωραία μέρη. Εστιάσαμε την προσοχή μας λόγω της κατάστασης αυτής. Κροατία, νέο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η κατάσταση με τους Σάμι στη Βόρεια Φιλανδία. Αυτοί ήταν οι λόγοι που μας οδήγησαν τις αποφάσεις μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. so, um, then I can... Uh, Προχωρούμε παρακάτω. Ελπίζω να ξεκαθάρισε η κατάσταση, τα πράγματα, τέλος πάντων. Στείλαμε και τις αποφάσεις των συντονιστών μετά τη συνεδρίαση του στις 19 Σεπτεμβρίου. Τώρα για τα διάφορα. Έχουμε τίποτε. Όχι. Οπότε θα ήθελα να ανακοινώσω ότι η επόμενη συνάντησή μας έχει προγραμματιστεί για τις 6 Νοεμβρίου από τις 9 το πρωί αλλά και το απόγευμα. Και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διερμηνείς και κηρύσω την λήξη της σημερινής μας συνεδρίαση. Ευχαριστώ.